στο διαδίκτυο, εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν έχει τον λόγο. Ο Επίτροπος, ο κύριος Στυλιανίδης. Καλημέρα σας, έχετε τον λόγο για να κάνετε την αρχή σας τοποθέτηση. Dear President. Ο κύριος Στυλιανίδης. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Συνάδελφοι, η σεξουαλική κακοποίηση των ε, παιδιών είναι ένα έγκλημα τερατώδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει δράση ούτως ώστε να καταπομίσει το φαινόμενο αυτό στο Ιντερνετ και εκτός του Ιντερνετ όσον αφορά αυτή την ε, οδηγία η οποία περιέχει διάφορα μέσα ούτως ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της απόκρισης των κρατών μελών όσον αφορά αυτά τα εγκλήματα. Και κατά αυτόν τον τρόπο επίσης θα διευκολυνθεί η διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κάποια τροποποίηση αυτής της οδηγίας στο εγγύς μέλλον. Θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην υλοποίηση αυτής. Οπότε και πρόκειται να δούμε πώς θα μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών αυτή η οδηγία. Τα δε αποτελέσματα πρόκειται τον Απρίλιο να δημοσιοποιηθούν. Κατόπιν θα έχουμε λήψη αποφάσεων όσον αφορά τις ε, παραβιάσεις που θα υπάρχουν και μεταξύ είμαστε σε διμερείς επαφές με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς αυτή η μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο θα βελτιωθεί και γίνονται σχετικές κοινοποιήσεις. Επίσης έχουμε κάποια ζητήματα συγκεκριμένα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου και το πώς οι δικαστικές αρχές μπορούν να αποσπάσουν κριτικά στοιχεία για τέτοιες περιπτώσεις κακοποίηση στο διαδίκτυο που βρίσκονται στα χέρια ε, νομικών προσώπων του τομέα και αυτό σε διαφορετικές ε, χώρες μέλη. Κάτι το οποίο αποτελεί έναν φραγμό ώστε να έχουμε αποτελεσματική έρευνα και δίωξη αυτών των εγκλημάτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν, θα πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων. Πρόκειται για κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν διάφορα κυβερνοεγκλήματα, διάφορα εγκλήματα τα οποία τα βοηθά το διαδίκτυο. Και ακριβώς επειδή το ίντερνετ πάει παντού σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε υπόψη το ότι χρειάζεται συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται επομένως μια συνολική προσέγγιση και έτσι να έχουμε μια συνέπεια. Επίσης, κατά αυτόν τον τρόπο να γίνεται η καταπολέμηση του εγκλήματος η κυβερνό ασφάλεια, η προστασία του καταναλωτή, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των δεδομένων αλλά και σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις προκλήσεις ως τμήμα του προβληματισμού μας για το επερχόμενο πακέτο μέτρων για τα ψηφιακά. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται στον την Παγκόσμια Συμμαχία κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στο διαδίκτυο. Πρόκειται για Παγκόσμια Συμμαχία και πρόκειται για δέσμευση πολιτική υπουργών από 54 χώρες οι οποίοι πρόκειται να λάβουν δραση δράση ούτως ώστε πρώτα-πρώτα να υπάρχει εντοπισμός αλλά και βοήθεια των θυμάτων να βελτιωθεί η ποινική δίωξη αλλά και η έρευνα να βελτιωθεί η συνειδητοποίηση και όπως να περιοριστεί η διάθεση στο διαδίκτυο αποτύπωσης της σεξουαλής κατοποίησης των παιδιών και αυτή η συμμαχία έχει αποδώσει σε πολλά μέτωπα. Οι δε δεσμεύσεις αποτελούν πλέον πολιτική μας. Ακόμη πάντως θα πρέπει αυτή η Παγκοσμία Συμμαχία να ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα πρώτα-πρώτα. Να εξασφαλίσει το ότι όλες οι χώρες θα συνεχίσουν την επιδίωξη των στόχων της πολιτικής μας με κοινέ προσπάθειες, επιστατεύοντας κοινού πόρους. Επίσης θα πρέπει να αγγίξει αυτή η συμμαχία περισσότερες χώρες. Θα πρέπει να αντιδράσει επίσης όσον αφορά τις απειλές, εκείνες που προκύπτουν στον πραγματικό κόσμο, ούτω ώστε η απόκριση να προσαρμοστεί σε ό,τι χρειάζεται. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε στενότερη συνεργασία με την βιομηχανία του διαδικτύου που έχει ρόλο να διαδραματίσει στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας. Και όσον αφορά το εσωτερικό Ταμείο Ασφάλειας, εμείς θα ξεκινήσουμε εταιρικέ σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για κάποιους πάρα πολύ σημαντικούς εμπλεκομένους. Αλλά και από την άλλη μεριά με αυτούς θα συνεργαστούν και οι αρχές. Και με την ε, με το Connecting Europe, αυτή την διευκόλυνση, θα ξεκινήσουμε αυτό το δίκτυο που αφορά το ίντερνετ και έτσι θα υπάρχει περισσότερη συνειδητοποίηση όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας για την προστασία των παιδιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτού του είδους τα κέντρα ε, του ίντερνετ ήδη λειτουργούν σε 27 χώρες μέλη όσον αφορά πρώτα-πρώτα κάποιο κέντρο, ούτως ώστε τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι να χρησιμοποιούν ε, όσο καλύτερα γίνεται το ίντερνετ. Δεύτερον, να έχουμε ε, κάποια κέντρα υποβοήθησης της εξοικείωσης με τα ψηφιακά, οπότε και θα υπάρξει και συνεργασία και με τη βιομηχανία αλλά και με τα σχολεία. Επίσης θα έχουμε κάποιο είδους ε, κέντρα βοηθείας, ούτως ώστε να συμβουλεύουν τα παιδιά και τα παιδιά να μάθουν πώς μπορούν να αναφέρουν οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά. Επίσης κάποια τηλεφωνική γραμμή για λήψη πληροφοριών που έχουν σχέση με παιδική πορνογραφία. Θα γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση όσον αφορά ε, το περιεχόμενο του ίντερνετ, και εάν χρειαστεί θα κοινοποιούνται τα επιλήφθηνα στοιχεία στις διοικητικές αρχές. Έτσι θα ελέγχονται οι πάροχοι του ίντερνετ. Και αυτό θα γίνονται με κάποιο μέσο πολιτικής το οποίο θα το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εφαρμογή του νόμου, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο εντοπισμό των ε, θυμάτων αλλά και των εγκληματιών. Και έτσι θα συγχρηματοδοτήσουμε το πώς θα έχουμε κάποιες κοινέ βάσεις δεδομένων που τώρα τις έχει η Interpol. Και έτσι η εφαρμογή του δικαίου και η επιβολή του νόμου θα γίνεται καλύτερη και θα γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις ομάδες τώρα το ΕΛΚ. Η κυρία Μόνικα Χόλμαερ για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για αυτή την ουσιαστική συζήτηση. Τελευταία έχουμε μια έκρηξη του αριθμού των πράξεων αυτών το ίντερνετ είναι ευλογία για πάρα πολλούς ε, τομείς ε, της οικονομίας αλλά και κατάρα για τα θύματα των εγκλημάτων. Έχω τις εξής ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Συστήσαμε το EC3 και ξέρουμε πως η βασική πλατφόρμα είναι το ίντερνετ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει επαρκές προσωπικό για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητας. Έχουμε όμως, μαθαίνω, τρία άτομα για ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως η Europol έχει ε, αρκετό προσωπικό, αλλά πρέπει να ασχοληθεί με την εμπορία ανθρώπων, με το οργανωμένο έγκλημα, με διάφορα πράγματα. Οπότε χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα ε, επαρκή στελέχωση. Δεύτερον, η εφαρμογή της οδηγίας που πρέπει να επιταχυνθεί στα κράτη-μέλη είναι μια οδηγία 2011, είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να εφαρμοστεί. Τρίτον, ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι εξαιρετικές και πρέπει να προωθηθούν. Τέτα, τελευταίον, πρέπει να εγγυηθούμε αφενός ε, την ιδιωτική ζωή αλλά όχι να προστατεύουμε τους εγκληματίες που βιάζουν χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Καπίνη. Τη δέχεστε. Η κυρία Καμπίνη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα αυτό. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση και τα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν με τα παιδιά. Όλα αυτά μας κάνουν να σκεφτούμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Χολμάιερ το εξή. Υπάρχει μια οργάνωση που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, ακούσαμε γι' αυτό. Η οργάνωση αυτή λοιπόν δίνει κάποια διασφάλιση για την προστασία του ιδιωτικού βίου γιατί προφανώς χειρίζεται στοιχεία από το διαδίκτυο. Πιστεύετε ότι ο οργάνωση αυτή που ανέφερε η Επιτροπή θα προσφέρει την εξασφάλιση αυτή για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Όταν γίνεται έρευνα σε δεδομένα ιδιωτικών εταιριών δεν γίνεται ατομικά και από ανθρώπους αλλά μέσω αλγορίθμων και μόνο όταν βρεθούν τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε τότε μπαίνει και ψάχνει ένα άτομο. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι σημαντική αυτή η αλγόριθμη και τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλδημοκράτες Ζίπελ για ένα... δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι πως πρόκειται για εγκλήματα, βαριά εγκλήματα που αφήνουν σωματικές και βαθιές ψυχολογικές πληγές. Και μέσω του διαδικτύου βεβαίως εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης έρχονται και σε επαφή με παιδιά οι δράστες μέσω του διαδικτύου. Το 2011 λοιπόν εγκρίναμε μαζί όλη μια οδηγία για να μπορούν τα κράτη-μέλη να αμυνθούν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο με κοινούς κανόνες, προδιαγραφές, ορισμούς των εγκλημάτων και ενιαίες διατάξεις για τις πινές, ακόμα και για εγκλήματα που γίνονται στο εξωτερικό. Η πρόληψη και η προστασία παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως και η βελτίωση βεβαίως της αντίληψης που έχουμε για το ίντερνετ. Βεβαίως, η απαγόρευση διαφόρων site είναι μόνο μεταβατική λύση θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική διαγραφή του περιεχομένου και εδώ πέρα δεν μπορούν να αποφασίζουν μόνο οι ιδιώτες. Ο λόγος για τον οποίο δεν εφαρμόζεται η οδηγία, από ό,τι φαίνεται, είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Το 2014 η Κομισιόν απίφθινε επιστολή σε 11, 11 κράτη-μέλη ότι θα κινήσει την διαδικασία επί παραβάση. Μόνο στην περίπτωση της Κύπρου δε ανεστάλλει η διαδικασία. Τα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη επιτέλους να κάνουν την δουλειά τους και η Κομισιόν θα πρέπει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της χωρίς να συγκρατείται στον τομέα αυτόν. Μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει λοιπόν να υποβάλει ένα σχέδιο οδηγία και αναμένω να δω πώ θα έχει αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξή. Η κακοποίηση δεν είναι εικονική. Λαμβάνει όντως χώρα στον πραγματικό κόσμο. Και δεν είναι δυνατόν να το αγνοούμε αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ έχετε ερώτηση από την ε, κυρία Χολμαϊρ, την οποία θα εγκρίνω κατ' εξαίρεση, γιατί μπλε κάρτα εγκρίνουμε όταν δεν μιλάει κανείς, ε, δεν έχει λάβει ήδη το λόγο. Δεν ήταν ανάγκη καν, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σίπελε αν ε, σοβαρά θεωρεί πως... Ε, το Google πραγματικά δεν, αν ανακαλύψει τυχαία ξέρω εγώ, τέτοιο υλικό, δεν θα πρέπει να το σβήσει αυτομάτως, αλλά να περιμένει τις αρχές. Το, το λέτε σοβαρά αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Νομίζω και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να δρουν. Εδώ, ε, δηλαδή όταν φτάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε πλέον για δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Απάντηση. Κυρία Χολμάιερ, ο κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος όταν πέφτει τυχαία πάνω σε ένα έγκλημα να παρεμβαίνει αλλά στην συζήτηση αυτής της οδηγίας παρατηρήσαμε πως υπάρχουν πέραν από τις αφείς περιπτώσεις και κάποιες οι οποίες είναι κάπως αμφίβολες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσφεύγει κανείς τις αρχές. Ευχαριστώ. Για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς, Τίμωθη Κέρκο, πια ένα λεπτό. Πρόεδρε, πώς προστατεύεται κάποιος σε μια κοινωνία. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει το απόλυτα σωστό και το απόλυτα άδικο. Δεν πρέπει να υπάρχει όμως σύγχυση. Εδώ πρόκειται για το χειρότερο των εγκλημάτων και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, για να τιμωρούνται οι εγκληματίες. Τα επιχειρήματα για ελεύθερη έκφραση κτλ. δεν έχουν νόημα εδώ. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε την κατάχρηση. Και η απάντηση είναι οτιδήποτε περνάει από το χέρι μα. Πρέπει να συνεργαστούμε με του παρόχου, με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, με τα σχολεία, με τι αστυνομικέ αρχέ κλπ. Πρέπει να σταματάμε κάθε τέτοια περίπτωση κακοποίηση στο διαδίκτυο. Πρέπει να διώκουμε, να συλλαμβάνουμε και να διώκουμε του εγκληματίε και να έχουμε στη διάθεσή μα ό,τι μέσο χρειαζόμαστε για το σκοπό αυτό. Πρέπει να νιώθουν ασφαλείς οι χρήστες του διαδικτύου. Και υπάρχουν και κάποια βασικά, Πρόεδρε, το διαδίκτυο φυσικά και το χρησιμοποιούμε όλοι, αλλά διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των φιλελεύθερων για δύο λεπτά η κυρία Γκρίσβεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από μερικές εβδομάδες στην Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη είχαμε μια συζήτηση με τους συναδέρφους ακριβώς για το θέμα του κυβερνοεγκλήματος και των κυβερνοεγκληματιών. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες φρικτές στατιστικές, στατιστικά δεδομένα, δηλαδή 4 εκατομμύρια υλικό πορνογραφικό βρίσκεται στο διαδίκτυο θύματα όλο και πιο μικρής ηλικίας. 10% είναι κάτω των 2 ετών. Εικόνες όλο και πιο βίες. Πρόκειται για ένα δίκτυο που κρυπτογραφεί με όλο και πιο περίπλοκο τρόπο κλπ. κλπ. Πριν από μερικές εβδομάδες, εγώ προσωπικά προσπάθησα, άρχισα να προσπαθώ να καταλαβαίνω πόσο λειτουργούν τα πράγματα σε αυτό το σκοτεινό δίκτυο. Και εκεί αντιλήφθηκα πόσο κρυφή πλευρά και σκοτεινή έχει το έγκλημα αυτό. Δυστυχώς οι κυβερνοεγκληματίες κάνουν κατάχρηση του διαδικτύου, κάτι το οποίο εμείς πρέπει να σταματήσουμε. Διαβάζοντας ε, επίσης τις σχετικές εκθέσεις, το 2014 διαπιστώσαμε μια αύξηση 100% για πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Διαπιστώσαμε δηλαδή για άλλη μια φορά ότι αυτή η παιδική πορνογραφία αυξάνεται στο διαδίκτυο περισσότερο από ποτέ. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτή η φρικαλαιότητα, στις δημοκρατίες μας, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, μπορούμε να έχουμε μια πραγματική έκθεση, μια πραγματική αξιολόγηση τι έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπενθυμίζω στην Επιτροπή ότι 13 Δεκεμβρίου του 2013 έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία αυτή. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει το ρόλο της που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Δεύτερον, τι γίνεται με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ε, Joint ε, Task Force της Europol για να αντιμετωπίζονται τέτοια κυβερνοκλίματα. Και τρίτον, κύριε Πίτροπε, δεν το αναφέρατε και λυπούμε γι' αυτό, πρέπει να καταργηθούν οι ιστότοποι και να μπλοκάρονται όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τέτοιες φρικαλαιότητες πορνογραφικού υλικού εκεί. Ευχαριστώ και περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό για τους αριστερούς η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως πρόταση βεβαίως ε, η καλή την οποία αναμένουμε είναι αυτή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Πρέπει να δούμε το ζήτημα από κάτω προς τα πάνω. Μόνο έτσι θα προστατευτούν τα παιδιά τα παιδιά κοβαλάνε τηλέφωνα στις ε, τσέπες τους και δεν ξέρουν τους κινδύνους ε, που σχετίζονται με αυτά. Πρέπει να δούμε λοιπόν την χρήση και τον κίνδυνο των νέων μέσων για να προστατεύονται τα παιδιά και να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί έχουν τρόπους ενημέρωσης. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε για το ίντερνετ. Ε, προσφάτως ε, στη δικιά μου την περιφέρεια, στη Βόρεια Ελλανδία κάποιες σχετικά αθώες ε, φωτογραφίες μαθητριών χρησιμοποιήθηκαν στο διαδίκτυο 732 τέτοιες φωτογραφίες μπήκαν σε πορνογραφικά site πράγματα που είναι σοκαριστικά απλά πρέπει να μάθουν τα παιδιά πόσο προσεκτικά πρέπει να είναι Άλλοι λένε πως αυτοί που τις ανέβασαν πρέπει να συλληφθούν. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος έχει τις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα και πως ε, ε, τις ανεβάζει κανείς νόμιμα ή παρανόμως. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους για δύο λεπτά, Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όλοι μας νομίζω θα πρέπει να χαιρετήσουμε την θεωρήση αυτής της ε, οδηγίας που θα συμβεί κάποια στιγμή φέτος και ότι είναι συγκλονιστικό το να ακούμε το πόσα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν ε, μεταφέρει στο ιστορικό δίκαιο τις ε, σχετικές διατάξεις γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το περιεχόμενο του ίντερνετ και στην οδηγία ξεκαθαρίζεται ακριβώς το ότι πρέπει να γίνει με τρόπο δεσμευτικό. Θα, τι θα πρέπει να μπλοκαριστεί θα, και θα πρέπει επίσης να ξεχαστεί το σχετικό δίκαιο το οποίο επίσης απαντά ένα ερώτημα που είχε ανακύψει προηγουμένως. Τι γίνεται δηλαδή με τους ε, παρόχους όπου και να βρίσκονται είναι ξεκάθαρο ότι η δράση πρέπει να αναλυφθεί, είναι ξεκάθαρο το τι ευθύνε έχει έκαστο σύμφωνα με την οδηγία. Μήπω θα μπορούσε να μα πει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει όσον αφορά το να τα συμφωνήσει με τι τρίτε χώρε, εκεί που πολλέ φορέ βρίσκονται οι πάροχοι, οι ιδιοκτήτε του τόσοι αυτών των ε, sites γιατί ε, αυτή η δραστηριότητα είναι απαράδεκτη όπου και να ε, εδράζεται. Επίση θα πρέπει να συνδέσουμε μεταξύ τους τις ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται όσον αφορά τα πιο ευάλωτα παιδιά, ας πούμε, τα μέτρα ούτως ώστε να ε, αναφέρεται ταχύως ποια παιδιά ε, έχουν χαθεί και επίσης θα πρέπει να υπάρχει για αυτά τα παιδιά ένα σύστημα εποπτείας ή παρακολούθησης. Είπαμε τώρα και για το σύστημα της πρόληψης θα πρέπει να υπάρχει για τους νέους, για τους ανήλικους γενικότερα ούτω ώστε οι ανήλικοι να ξέρουν και να αναγνωρίζουν τους κινδύνου. Είναι πολύ σημαντικά τα κέντρα που αναφέρθηκαν. Είναι και επίση σημείο επαφής για τα παιδιά που δεν μπορούν, ε, δεν θέλουν να αναφέρουν το τι γίνεται όσον αφορά του σχολείου, του γονεί του, να δούμε επίση αν υπάρχει κάποιο είδου εξωτερική διαπαιδαγώγηση, να ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ. Αναφέρατε ε, συνάδελφοι τα σχετικά με την ε, μεταφορά της ε, οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο θέμα για το οποίο πολλά κρατημέλη έχουν ε, βραδύνει πολύ αλλά θα πρέπει να δούμε και το ότι πολλές φορές έχουμε δυσκολίες να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και εκεί υπάρχουν φράγμοι πολύ. Εδώ είμαστε ομόφωνοι για το θέμα όμως τελικά. Για ποιο λόγο κάποιες κυβερνήσεις, κάποια κρατημέλη δεν κάνουν ό,τι πρέπει. Λάμπερτ. Νομίζω θα μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί αργούν κρατημέλη να εφαρμόσουν την οδηγία. Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις το θέμα είναι κατά πόσον κάτι είναι σύντονο με το ιστορικό δίκαιο, τι γίνεται με τις ποινές, αν είναι πιο βαριές, πιο ελαφρές που προβλέπονται αλλά και κάποια κρατημέλη όπως η δική σας χώρα ακόμα δεν έχουν απλώς ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Άρα θα πρέπει να απευθυνθούμε στους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων εκεί να τεθεί το θέμα του γιατί δεν έχει εφαρμοστεί η οδηγία. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Diane Dodds, μία γεγραμμένη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είναι το ίντερνετ μια γέφυρα για να δώσει ευκαιρίες σε καταναλωτές, σε επιχειρήσεις, αλλά επίσης από την άλλη μεριά δίνει ευκαιρίες και στους εγκληματίες που ενεργούν βάσει των παιδιών. Οπότε και εμεί θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, να βρούμε κάποιες λύσεις να καταπολεμήσουμε τέτοιε κακοποίησει. Στην ε, Βόρεια Είχαμε μια ανεξάρτητη μελέτη τον Νοέμβριο του 2014, την έκανε η Κάθλιν ε, Μάρσολ και κατέληξε στο ότι είχαν εντοπιστεί έξι ε, τέτοιες περιπτώσεις κακοποίησης στο διαδίκτυο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σε ένα σχολείο επίσης, ε, σε άλλη μια περίπτωση εντοπίστηκε το ότι η κακοποίηση είχαμε από το 2008 πέντε περιπτώσεις και 22 το 2014. Επομένως ε, διαπιστώθηκε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Είχαμε κάποιους 16χρονους οι οποίοι επίσης είχαν υποστεί τέτοια αποτρόπια κακοποίηση. Θα πρέπει, συνεχίζει η ομιλήτρια, να εξασφαλίσουμε το πώς τα παιδιά μας θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ αλλά επίσης να εξασφαλίσουμε για το ότι αυτοί οι γίγαντες οι οποίοι κυριαρχούν στο ίντερνετ διακόπτει ο πρόεδρος, κλείνει το μικρόφωνο λυπούμε αλλά κατά πολύ υπερεύεται το χρονικό όριο Ταντέος Διεύκα είναι ο επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε ναι, δεν έχω. Με πολλού τρόπου βλέπουμε ότι υπάρχουν εγκλήματα τα οποία διαπράττονται στο Ιντερνετ κατά κάποιων ανηλίκων και αυτά είναι πάρα πολύ συμβουλευτικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το, το, αρχίσαμε να συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το πρόβλημα και έχουμε κάποιες τέτοιες ε, διαδικασίες αλλά μόλι πολύ πρόσφατα και αυτό δεν είναι σωστό ε, έχουμε την Europol και η οποία μας λέει ότι έχει αυξηθεί αυτό το έγκλημα. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στην, στην, στην ε, αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος. Άρα θα πρέπει να δούμε το... τι πορεία θα πάρει η αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος. Γιατί θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε ε, κάποιες ε, τακτές επαφές με άλλα ε, κράτη να δούμε τι γίνεται εκεί που πηγαίνουν αυτοί οι εγκληματίες ας πούμε στα νησιά Καϊμάν και πώς κανείς θα μπορεί να καταγγείλει αυτού του είδους τα αποτρόπια σεξουαλικά εγκλήματα. Χρειάζεται επίσης περισσότερη εναρμόνιση, ούτως ώστε να μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτά τα εγκλήματα και επίσης να γίνει πιο εντατική η συνεργασία των ε, διοικητικών αρχών που καταπολεμούν αυτά τα εγκλήματα. Επομένως, εδώ το θέμα δεν είναι μόνο καταπολέμηση του εγκλήματος με καταστολή, αλλά χρειάζεται να γίνουν ενέργειες και μέσω της εκπαίδευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να τηρείτε το χρόνο σας, γιατί στις 11 θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Αν ο καθένα ξεπερνάει το χρόνο του, καταλαβαίνετε ότι δεν θα προλάβουν να μιλήσουν όλοι όσοι είναι γεγραμμένοι και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τι ψηφοφορίε στην γνώρα μα. Η κυρία Ντάλη, τώρα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφερόμαστε εδώ σε εκατομμύρια παιδιά που είναι θύματα της πορνογραφίας στο διαδίκτυο. 20% αφορά παιδιά κάτω των 10 ετών είναι αυτή η πραγματικότητα και είναι τρομερό έχουμε να κάνουμε με μια παράνομη δραστηριότητα η οποία καταστά πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που είναι θύματα. Εδώ μιλάω και ως εκπρόσωπος βέβαια του λαού αλλά και ως μητέρα. Ξέρω παιδιά που ήταν θύματα αυτού του εγκλήματο. Πρέπει να τα προστατεύουμε, να τους προσφέρουμε μια ειρηνική δουλειά, να μπορούν ελεύθερα να παίζουν με τα παιδιά τους και κανένας να μην τους κλέβει την αθωότητα. Το διαδίκτυο είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών, αλλά δυστυχώς μπορεί να έχει και σαν αποτέλεσμα πολλοί να κατεβάζουν πορνογραφικό υλικό με θύματα τα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να σταματάμε το διαδίκτυο, να το κόβουμε. Είναι αυτή η λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει νέες τεχνολογίες, όπως τα Darknet για παράδειγμα, που ανώνυμα ξέρουμε ότι ορισμένοι μπορούν να κατεβάσουν τέτοιο υλικό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα συζήτησαν τη διαδικασία ανώνυμους και θα έπρεπε τέτοιες προσπάθειες να τις επεκτείνουμε για να αποφύγουμε την παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει λοιπόν να προσαρμόσει την οδηγία της του 2011 και να λάβει υπόψη τη νέα αυτή πραγματικότητα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο ξέρετε ότι παραμένουν για όλη τη ζωή των παιδιών εκεί, στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε. Κύριο κρύπεκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χάρη στις νέες τεχνολογίες έχουμε μια νέα γενιά παιδιών που μεγαλώνει, που γνωρίζει την τεχνολογία αυτή καλύτερα από τους γονείς και τους δασκάλους. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά. Αλλά συχνά τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που τους απειλεί ε, στο διαδίκτυο όταν επικοινωνούν με κάποιους ή όταν μπαίνουν σε κάποιες ε, σελίδες. Ε, ως βουλευτής ήδη του Σλοβακικού Κοινοβουλίου είχα επισημάνει το πρόβλημα και η εκστρατεία μου είχε στόχο την ε, νομική προστασία των παιδιών από τέτοιο επικίνδυνο περιεχόμενο. Μαζέψαμε πάρα πολλές ε, υπογραφές ε, σε μια καμπάνια και είμαι πεπισμένος πως ο αγώνας αυτός ε, ξεκινάει οπωσδήποτε και στα ΜΜΕ και σε νομοθετικά βήματα. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών στο διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Τα παιδιά όλο και πιο μικρά και βεβαίως οι εικόνες αυτές κυκλοφορούν ε, σε όλο τον κόσμο σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το 2011 λάβαμε μια απόφαση να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό και τώρα η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει μια έκθεση και συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία θα έχουν νόημα. Η έκθεση δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία για αυτή την δουλειά. και πρέπει να είμαστε πράγματι προετοιμασμένοι για το μέλλον και θα πρέπει επιτέλους να πιάσει κομισιόν τον τάβρο από τα κέρατα. Πράγματι σας ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο. Ρόπε τώρα έχει τον λόγο. Ačiū Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να τα βάλει με αυτό το φοβερό έγκλημα. Το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, είναι γνωστό. Η επιβολή του νόμου δεν πετυχαίνει πάντα γιατί οι αρμόδιες αρχές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους το έγκλημα. Πρέπει όμως να αναλάβουμε την ευθύνη για τα εγκλήματα αυτά. Και ξέρουμε ότι οι αρμόδιες αρχές ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είναι καταρτισμένες οι αρχές κατάλληλα, οι αστυνομικοί κλπ. Οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Η πληροφόρηση πρέπει να φτάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως επίσης και οι αποδείξεις και πρέπει να αναβαθμίσουμε τα σχέδιά μας για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από την ε, κυρία Μουσολίνη. Τη δέχεστε? Κυρία Μουσολίνη. Θέλω κατά να σας πω για την ε, τελευταία παρέμβαση. Παρακαλώ, συνάδελφε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πώς μπορεί να είναι κοινοτικό δίκαιο το να διευκολυνθεί η καταγγελία και γιατί αυτό επιβάλλεται. Ε, αυτό θα είναι ένα καμπανάκι κινδύνου ούτω ώστε να παρωθεί κάποιον να το κάνει και να υπάρχει δυνατότητα για καταγγελία τέτοιου περιεχομένου πορνογραφικού στο ίντερνετ. Κύριε Ροπέ, σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την ερώτηση. Νομίζω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα με τρόπο βεβαίως οικονομικό και πρέπει να γίνει μια μελέτη νομίζω. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι πραγματικά ένα αειδιαστικό έγκλημα. Έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο που αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 80.000 περισσότερα αρχεία. Δεν σβήνουν αυτά τα αρχεία και η κατάσταση είναι δραματική. Η Μεγάλη Βρετανία ακολουθεί εδώ πέρα τη βέλτιστη πρακτική. Υπάρχει συγκεκριμένο αδίκημα ε, που αφορά την κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο. Υπάρχει ειδική μονάδα της ε, αστυνομίας ε, και των μυστικών υπηρεσιών που μπαίνει στο, σκοτικό, στο σκοτεινό δίκτυο και συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού και βεβαίω και 50 εκατομμύρια λίρες για το Ταμείο Προστασίας των Παιδιών. Δυστυχώς όμως ε, η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι σαν τους τρομοκράτες και ανάλογα πρέπει να συμπεριφερθούμε στο εθνικό και διεθνές επίπεδο και να εξοπλίσουμε ανάλογα τις αρχές. Ευχαριστώ. Όχι, με συγχωρείτε. Για 1,5 λεπτό. Δίας Δεμέρα Γκαρθία Κονσουέκρα. Ευχαριστώ. Πάνω από ένα εκατομμύριο πορνογραφικές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με θύματα τα παιδιά. 50.000 με 100.000 ε, παιδόφιλοι κυκλοφορούν εικόνες στο διαδίκτυο. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και η οδηγία πρέπει να ενημερωθεί και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να έχουμε κοινό στόχο με τη συμμετοχή των αστυνομικών και άλλων αρχών που πρέπει να διώκουν τους εγκληματίες. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν και εγγύσεις όσον αφορά την δίωξη των εγκλημάτων αυτών και όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων στα ποινικά δικαστήρια για να μην στιγματίζονται τα παιδιά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε τα σφάλματα. Άρα τεχνολογικές λύσεις. Είναι αναγκαίο το SRR να αντιμετωπιστεί και να εξαφανιστούν οι σελίδες με το πορνογραφικό υλικό, να αντιμετωπιστεί η διανομή τους μέσω ειδικών δικτύων peer-to-peer. Να υπάρχει και ένας κώδικας δοντολογίας όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και όλα αυτά με συντονισμό σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών. Είναι θέμα ασφάλειας πρέπει να συμμετέχουν αρχική κοινωνία των πολιτών να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της ε, Europol, της Eurojust και επίσης να δούμε τι γίνεται με την εμπορική εκμετάλλευση τέτοιου πορνογραφικού υλικού επίσης στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε μπλε κάρτα από την Μπόσαν. Θέλε, δέχεστε. Μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Ναι. Ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, αναφερθήκατε στη νομική προστασία και στη νομική προστασία. Όμως, χρειάζεται χρόνος για να εμπλακούν τα δικαστήρια. Μέχρι τότε θα έχουμε πολλά νέα θύματα. Η διαπαιδαγώγηση σεξουαλική δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική στα σχολεία. Τι λέτε γι' αυτό. Απάντηση. Αναμφίβολα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί ένα μέσο, αλλά όχι το μόνο. Φυσικά, αυτό που χρειάζεται είναι να καταδικάζονται οι εγκληματίες. Δυστυχώς, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι προστατεύεται περισσότερο εγκληματίας παρά το θύμα. Κάθε νομοθετική αστυνομική διάταξη πρέπει να έχει σαν στόχο να προστατεύει τα θύματα. Γιατί αυτά τα θύματα είναι ειδικά θύματα, είναι παιδιά, άρα αξίζουν τη μεγαλύτερη δυνατόν προστασία. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, περνάμε τώρα στη διαδικασία HDI. Έχω ένα κατάλογο ο είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις ε, συνήθεις οπότε δεν θα μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω λίγο να τα μοιράσω κάπως δίκαια η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Λεσάνες. Πρόεδρε, χάσαμε πολύ χρόνο. Τόσα χρόνια έχουν περάσει χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη έκθεση. Οπότε θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να κάνουμε τον κόδωμα. Αλλιώ θα χάσουμε αυτή τη ε, μάχη. Γιατί όπω ξέρετε, στη σκοτεινή πλευρά του Ιντερνετ όλα προχωράνε όλο ένα και πιο γρήγορα. Οπότε θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τι γίνεται. Όπω είπατε, ε, αναχώρα και τελικά θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και τα παιδιά αλλά και τους ε, γονείς αλλά και τους δασκάλους και επίσης να υπάρχει μια ανοιχτή πράσινη γραμμή ε, πανευρωπαϊκή για αυτό το θέμα και επίσης να φιλτράρουμε, να μπλοκάρουμε κάποια website γιατί τελικά από ό,τι φαίνεται η Europol δεν κάνει αρκετά. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε ούτω ώστε να μπορεί καλύτερα να ερευνήσει, να βρει του εγκληματίε, να εντοπίσει επίση και τα θύματα και έτσι να είναι ευκολότερη η ανταλλαγή των δεδομένων, να προστατεύσουμε τα παιδιά μα. Άρα χρειάζεται μια τέτοια κινητοποίηση και αυτό πρέπει να γίνει και από εμά του πολιτικού αλλά και από όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρίτσαρτ Χάουιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα την ε, ημέρα του πιο ασφαλούς ε, διαδικτύου χαίρομαι που κάνουμε αυτή την συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε το κατέβασμα τέτοιων αρχείων και να διώκονται οι χρήστες όπου και αν βρίσκονται στον ε, κόσμο. Πέρσι η σχετική υπηρεσία κατέβασε πάνω από 30.000 αρχεία από το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν ε, ακόμα υποθέσεις της δεκαετίας του 1970 που εκδικάζονται. Υπάρχει, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές υποθέσεις ε, για κακοποίηση και προετοιμασία παιδιών για κακοποίηση. Πρέπει λοιπόν εμείς να δώσουμε τα εργαλεία στις διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Μιχαέλα Σόλτοβα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Θέλω να σας ευχαριστήσω. Προσωπικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες οι χώρες μέλη πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό στο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε σε πολλές δυνατότητες ε, στην εφαρμογή της οδηγίας του 2011, για παράδειγμα, αλλά θα ήθελα μια λεπτομερή αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Γιατί δεν προτείνουμε νέα αρρύθμιση, δεν προτείνουμε νέα οδηγία, όμως θα θέλαμε να γνωρίζουμε η οδηγία που έχουμε σήμερα πώς αποτελεσματική είναι, πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα, δεδομένου ότι έχουμε όλο και περισσότερα θύματα. Προφανώς όλα αυτά τα νομοθετικά μέτρα δεν επαρκούν ή δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Είναι μέτρα τα οποία δεν φτάνουν και τελικά δεν καταφέρουν να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς τους εγκληματίες. Δηλαδή η απάντησή σας ποια είναι για να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και πώς θα έχουμε καλύτερα συνειδητοποίηση από πλευρά των παιδιών, των γονιών και των σχολείων. Ευχαριστώ η κυρία Τόμασετς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το Υπουργείο στην Κροατία το 2013 έκανε μία έρευνα και είπε ότι κάθε πέντε παιδιά ένα έχει προβλήματα στο διαδίκτυο και ένα 30% έχει εκτεθεί κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Οι υπεύθυνοι βέβαια σήμερα κρύβονται πίσω από ένα ψεύτο προφίλ στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι γονείς και τα παιδιά να είναι πιο συνδυτοποιημένοι, να μην περιμένουν να γίνουν θύματα, αλλά να προλαμβάνουν την κατάσταση αυτή. Πρέπει να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους και όχι να γίνονται θύματα επικοινωνώντας με άγνωστους στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να το προλαβαίνουμε. Να υπάρχει δηλαδή κάποιο είδου κόκκινο κουμπί και να ενισχύσουμε όλη τη λογιστική που βρίσκεται πίσω από τα δίκτυα αυτά. Ευχαριστώ για ένα λεπτό συνάδελφο συνάδελφος Ιγνάσιο Κοράο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Μιλάμε εδώ πέρα για το ευρώ, μιλάμε για άλλα θέματα, αλλά όμως τώρα πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί κάποια λύση γι' αυτό. Να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, γιατί ξέρουμε τα θετικά του ίντερνετ, γιατί από τη μία μεριά έχουμε ένα μέσον το οποίο μας βοηθά να ερχόμαστε κοντά, να βρίσκουμε ό,τι να είναι. Αλλά από την άλλη μεριά ε, έχουμε την σκοτεινή πλευρά. Έχουμε εκεί πέρα αυτά τα εγκλήματα που εκφεύγουν του ελέγχου μας. Πολύ σοβαρά εγκλήματα αφορούν ακόμα και ανήλικους κάθε ηλικία ακόμα και δύο ετών. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις ενεργέ μας γιατί πάρα πολύ γρήγορα εξελίσσεται το ίντερνετ και έτσι να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ κύριε Κοράου. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Ζαμπόρσκα για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Να ευχαριστήσω την Μόνικα Χολμάιερ για το ότι επισήμανε το θέμα της επικαιροποίησης και εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Και συμφωνώ και με το αίτημα η Κομισιό να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης ε, για να βοηθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα τους κινδύνους του διαδικτύου στη Σλοβακία υπήρχε μια τέτοια καμπάνια με τίτλο «Ξέρετε τι κάνει το παιδί σας». Και βεβαίως ε, πρέπει να ενημερώσουμε και για τους κινδύνους, όπως ενημερώνουμε για τους κινδύνους του αλκοόλ ε, και διαφόρων άλλων πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να γίνει προτεραιότητα της Ένωσης ε, και να αφιερώσουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Ευχαριστώ ακριβώς ένα λεπτό και δίνω τον λόγο ξανά στην Κομισιόν. Κύριε Στυλιανίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας σήμερα αυτή την πρόκληση και αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει βήματα για να αντιμετωπίσει την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Δυστυχώς όμως, ο αγώνας αυτός, η μάχη για την κατάργηση αυτού του απεχθούς εγκλήματος, δυστυχώς δεν έχει ακόμα κερδιθεί. Δυστυχώς. Συνεπώς πρέπει να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε μια πολιτική η οποία να σέβεται και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πολιτών, να διασφαλίζεται την αποτελεσματική διαρεύνηση και δίωξη τέτοιων εγκλημάτων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και να διασφαλίζονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Όμως, πράγματι, όπως είπαν και η Μόνικα και άλλοι, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό στα διάφορα κέντρα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ενίσχυση της Europol. Είναι ζωτική σημασία. Το αναγνωρίζουμε, νομίζω αυτό, όλοι αυτή την ανάγκη. Όμως θέλω να επαναλάβω κιόλα ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας λοιπόν για να ενισχύσουμε τη συνειδητοποίηση του κόσμου σε αυτό το θέμα όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τελείωσε άρα η συζήτηση για αυτό το θέμα.